Ε, η θητεία του κυρίου Γιώχανσον. Ο κύριος Ελί Χοουραό μου ανέφερε ότι παρετείται από Ευρωβουλευτής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 1 και 3 το Κοινοβούλιο το σημειώνει και θεωρεί ότι χειρεύει ε, η θέση του από την 4η Ιανουαρίου 2012. Ο πρόεδρος του